Madame le Président. Bonjour à tous. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όσους είναι παρόντες. Άρχεται η Σύνοδο. Η η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κέντρα επιχειρήσεων στην Ασία. Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη τη προφορική ερώτηση, τον κύριο Μορέιρα δηλαδή, για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,